I would like to ask everyone to sit down. Η κυρία Κίνγκα Γκόντς, σας παρακαλώ να καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία που προβλέπεται μακροσκελέστατη. we would like Ας καλωσορίσουμε πρώτα τα μέλη της Επιτροπής ε, Οικονομικών καθώς και βεβαίως τα μέλη μας της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών καθώς και το προσωπικό των επιτροπών αυτών. Μάλιστα, εσείς. Ο κ. Γκοζές να επισημάνω μόνο στους συναδέλφους μου του Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής ΕΚΟΝ ότι θα πρέπει να παρακολουθούν τι κάνει ο συνάδελφός μας Κάρινς που κάθεται εδώ μπροστά μου. Α, πολύ σημαντική πληροφορία, λέει η κυρία Γκόντς. Πριν αρχίσουμε όμως πραγματικά την ε, ψηφοφορία, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με δύο διορθώσεις. Παρακαλώ ακούστε γιατί είναι σημαντικές. Ε, πρόκειται για δύο διορθώσεις στην λίστα ψηφοφορίας όπως αυτή κυκλοφόρησε χθε το βράδυ. Η μία αναφέρεται στη συμβαστική Β. Η δεύτερη προφορική τροπολογία της ΓΚΟΕ για τα ποσοστά, 10% λέει εδώ, έχει ζητηθεί και από τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Εάν γίνει ε, δεκτή η προφορική τροπολογία, τότε οι τροπολογίες 214, 15, 220 και 21 εκπίπτουν ως συνέπεια αυτού ή καταπίπτουν. Μπορέσατε να παρακολουθήσετε αυτό που είπα. Το άλλο είναι πάλι στην Β τροπολογία προφορική της Άλντε για την επέκταση και σε άλλα μέλη των οικογενειών. Θα υπάρξει και τρίτο, όπου λάθος αναφέρεται στο ΤΕΒΕ 13. Τα λέω αυτά βέβαια ιδίως για εκείνους που θα υποδεικνύουν πώς να ψηφίζουν οι διάφορες πολιτικές ομάδες. Αν μπορέσατε να παρακολουθήσετε... Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, συνεχίζει η κυρία Γκόνς, είναι να κάνουμε πρώτα μια ενδεικτική ηλεκτρονική ψηφοφορία πριν αρχίσουμε, γιατί είναι τόσα πολλά τα μέλη. Ας κάνουμε μια δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, δοκιμαστική, αρχίζει. Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα. Ήταν λοιπόν πολύ ορθή η συμβουλή να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί η κάρτα μου, λέει κάποιο. Φαίνεται πως δεν λειτουργεί ολόκληρο το σύστημα, λέει η κυρία Γκόνς. Θα χρειαστούμε λοιπόν κάποια τεχνική υποστήριξη και θα δούμε μετά αν λειτουργούν οι διάφορες κάρτες ή όχι. Ας δοκιμάσουμε ξανά. όχι ακόμη δεν είναι το σύστημα παρακαλούμε να παρέμβει ο τεχνικός. Please you've got arrows on. I haven't even got arrows. Do we Please wait a minute. The technician is coming and hopefully we're correct. Περιμένετε λίγο. Έρχεται ο τεχνικός. Και μετά θα ελέγξουμε και τις κάρτες. It is not recognizing any of the cards. Earlier it recognized the Libra cards and not. Δεν αναγνωρίζει καμία κάρτα το σύστημα από τι φαίνεται. We are really sorry we had a vote before. Λυπούμεθα. Κάναμε ψηφοφορίες το πρωί και πήγαν μια χαρά. Πρόεδρε, νομίζω ότι η βιομηχανία των χαρτοπαιχνίων, των παιχνίων γενικότερα έχει κάνει παρεμβάσει στο σύστημα ψηφοφορίας. Βλέπετε πώς δουλεύουν τα λόμπι πια. Ε, μπορεί να έχουμε πολλές συνομωτικές θεωρίες για να εξηγήσουμε την κατάσταση. Ελπίζουμε όμως το σύστημα να δουλέψει. Το σύστημά μου λέει ότι πρέπει να γυρίσω την κάρτα ανάποδα. Then I think all of the conspiracy theories might be valid. But you know that Libe is is the committee dealing with conspiracies, different conspiracies. Γενικά η Λίμπε ασχολείται με τις συνωμοσίες. Και σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο κλίμα εργασίας μας.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 θα ήθελα λίγη υπομονή από πλευρά σας, θα μας πούνε αν μπορούν να διορθώσουν το σύστημα, αλλιώς θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το τι θα κάνουμε. Τώρα μόλις μου είπαν ότι ξαναρχίζει εκ νέου το σύστημα να δουλέψει και αυτό απαιτεί πέντε λεπτά. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλα πέντε λεπτά για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. μιλήστε μεταξύ σας, κάντε παρέα. Or restart it, then we can start the vote. Thank you. Now, uh, Ας κάνουμε τώρα την δοκιμαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελπίζω να ε, έχει θετική, να έχει αίσια έκβαση δηλαδή. Αρχίζει τώρα η δοκιμαστική ψηφοφορία. Κάποιες θετικές ψήφοι φαίνεται να λείπουν. Έξι. Τώρα ε, ελέγξτε τις κάρτες σας. Yeah, no, eh, two is, is still missing. One is missing. Push more your Πατήστε καλά, βάλτε καλά τις κάρτες σας μέσα και πατήστε καλά το κουμπί. Μία μας λείπει ακόμα. Ελέγξατε την κάρτα σας καθώς και την ψήφο που δώσατε. Λίγη ψηφοφορία εδώ. Είναι εντάξει λοιπόν. Πολύ καλά. Τότε μπορούμε να αρχίσουμε. Και ας τώρα αποτελεσματικές και αποτελεσματικοί. Συμβαστική, συμβαστική μείον αλφα. Εδώ οι πράσινοι έχουν ζητήσει κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά, λέει η πρόεδρος. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη. 35 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική Α Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τμήμα τρίτο. Υπέρ, κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λήξη. 32 υπέρ, 30 κατά. Εγκρίνεται. Τμήμα τέταρτο. Κατά. Αποχές. Τμήμα τέταρτο. Υπέρ. Τμήμα τέταρτο πάλι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Πέρας. Ε, 36 υπέρ. Να σηκώνετε καλά τα χέρια σας. Ακολουθεί 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 187. Όχι, 188. Υπέρ. 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Διακόσια ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. δύο υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, 202. 30 υπέρ 33 κατά απορρίπτεται. Τρεις προφορικές τροπολογίες. Κατά παράδοση η Econ Committee αρχίζει πάντα με τις προφορικές. Πρώτη. Ποιος υποστηρίζει. Κατά. Αποχές. Θα χρειαστεί παρήθευση. Λήξη ...27 υπέρ, 36 κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερη προφορική τροπολογία... ...της ΓΚΟΕ και των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών. Ποιος την υποστηρίζει υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3 της Άλντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Συμβαστική 3. Ίσως είπε C η πρόεδρος. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ορισμένες τώρα εκπίπτουν γυρίζω δύο σελίδες και πηγαίνω στην 225 Όλες οι άλλες οι εκπίπτουν. Και τώρα έχω την 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Διακόσιες, 200 μάλλον 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή επαλήθευση 25 υπέρ, 38 κατά. Απορρίφθηκε λοιπόν και με διαφορά. Συμβαστική σε γάμα δηλαδή. Υπέρ, Μια στιγμή να ελέγξουμε. Συμβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική D, δέλτα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική ε. Αρχίζουμε πάλι με τις προφορικές τροπολογίες. Τμήμα πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε, αλλά πάντως απερίφθη σαφώς. Λήξη. 23 υπέρ, 39 κατά. Προφορική τροπολογία 2, λέει ο τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλά λοιπόν, ολόκληρη τώρα η συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, σιγματάφη δηλαδή. Υπάρχουν πολλές που εκπίπτουν στο μεταξύ. όπως Φόξτροτ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται αυτή. Και προχωρώ στην 271, υπέρ, κατά, αποχές, αυτή απορρίπτεται. Επαλήθευση, καλά. 271 επαλήθευση. Απορρίπτεται, αλλά με ισοψηφία. Συμβαστική G, Golf, άρθρο 8, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283 δεύτερο μέρος υπέρ υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε να επαληθεύσουμε Μάλιστα. Ω, βεβαίως, απορρίφθηκε, σαφώς. 285, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 287, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική age. Ήτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I. Ιώτα. Άρθρο 10. Αρχίζουμε πάλι με την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ζητείτε δε και ψηφοφορία κατά τμήματα σε δύο μέρη, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Συμβαστική J. Με την προφορική τροπολογία πάλι, ψήφι υπέρ, Και Απορρίπτεται. Α, θέλετε επαλήθευση. Ψηφίσατε την 301 ή απλώς την επιδείξατε. Στη δική μου, λέει η πρόεδρος λίστα, λέει ότι είναι εγκεκριμένη. False if compromise I is adopted, λέει. Εκπίπτει επομένως. Έχουμε τώρα το J και προφορική τροπολογία πάλι. Αρχίζει η επαλήθευση μιας και τη ζητήσατε. Λήξη. 33 υπέρ και 27 κατά. Δεύτερη προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Προφορική τροπολογία 2. Λήξη. Πού βρισκόμαστε. Είστε όμως σίγουροι όλοι. Είμαστε στη συμβαστική τροπολογία J. Και επειδή βασιζόμαστε στις παραδόσεις της Οικονομικής Επιτροπής, γι' αυτό αρχίζουμε με τις προφορικές τροπολογίες. Πρώτα ψηφίζουμε λοιπόν τις προφορικές τροπολογίες και τώρα έχουμε φτάσει στην δεύτερη προφορική τροπολογία πριν να ψηφίσουμε την ε, συμβιβαστική. Και ίσως το πρόβλημα να είναι, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις διάφορες ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Αρχίζουμε τώρα εμεί σε όλε τι ψηφοφορίε με τι προφορικέ τροπολογίε. Και όταν θα έχουμε ξεκαθαρίσει την άποψή μα για τι προφορικέ τροπολογίε, τότε θα ψηφίσουμε την συμβιβαστική. Ψηφίσουμε τώρα την δεύτερη προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει δεύτερη προφορική τροπολογία στη δική μας λίστα, λέει ο κ. Κίρκ Χόπ. Μα υπάρχει και στη δική σας λίστα. Η πρώτη να μου επιτρέψετε να διαβάσω το κείμενο. Τη δεύτερη λέει τώρα. Απορρίφθηκε. Βρήκατε τη δεύτερη τώρα. Α, ωραία, ναι, ναι. Πρέπει βέβαια να προσαρμοστούμε στο διαφορετικό σύστημα. Παρακολουθούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Ωραία. Είμαστε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία κατά τμήματα στην συμβαστική τροπολογία. Στο πρώτο μέρος λέει η πρόεδρος τώρα. Ε, υπέρ. Τώρα μετά από τις προφορικές τροπολογίες ψηφίζουμε την συμβαστική. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε ναι. Ψηφίσαμε τις δύο προφορικές τροπολογίες, τώρα ψηφίζουμε την συμβιβαστική τροπολογία σε δύο μέρη. Και τώρα μιλούμε για το πρώτο μέρος, για το πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Πρώτο τμήμα της, προφορικής, της ε, τροπολογίας. Πρώτο τμήμα της συμβαστικής. Κατά, αποχές, εγκρίνεται σαφώς. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτό. Τώρα συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική λάμδα, έλα, αγγλικό. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της L. No, it, it Compromise L, uh, second part. Λοιπόν ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της L, λάμδα. No. <laughs> Okay. Uh, electronic vote is closed. Τέλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. <laughs> Okay, uh, uh, the vote is closed. Yeah, it is 34 uh, plus and 28 minus. It is adopted. Uh, the next one is... Επόμενη, η 321 ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική M, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία. 329 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Don't confuse people more. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. νη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 339. τριάντα Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 340 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τζούρι 23 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μαζί με τη 225 λέει πρόεδρος, την ψηφίσαμε. Η επόμενη λοιπόν, 352, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 352. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική ο όμικρον. Υπάρχει μια προφορική εδώ. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η προφορική. Υπάρχει τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 244 δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 58 ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή 59 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική π αγγλικά ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική Q εννοεί η πρόοδος. Και εδώ έχουμε προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας στην Q. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα η συμβιβαστική Q. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4.24. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή. But it, is, it was clearly adopted. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. 39 plus and 21 minus is clearly adopted. 39 υπέρ 21 κατά. Γίνεται δεκτή. 28. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική R αγγλική. είναι υπέρ. Για μια στιγμή. Έπρεπε να ψηφίσουμε την 154. Εκατόν πενήντα τέσσερα έπρεπε να την ψηφίσουμε.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 με διαφορετικό αριθμό σελίδας. Άρθρο 27. Νέο. 154. Ο αριθμός τροπολογίας. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σαφές. Ευχαριστώ που μας το υπενθυμίσατε. Συμβιβαστική R. Ρο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τέσσερα και 4.45 από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 4.44 και 4.45. Τέλος. Απερίφθη. Τετρακόσια πενήντα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 450. Τέλος.

78 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εβδομήντα εννέα και 35 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές 453 υπέρ κατά Αποχές. Απερίφθη. 400... Α, για μια στιγμή. 454. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 455 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 455. δεκτή. Συμβιβαστική S. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τέσσερα εξήντα πέντε. Ποιοι είναι υπέρ. Και τέσσερα εξήντα έξι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 467 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 467. Τέλος. Δεκτή. Παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας ψηλά. 468 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 468 ελέγχουμε. Τέλος. 30 υπέρ 28 κατά δεκτή. 469 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 470 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 470. Τέλος. Απορρίπτεται. 471 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 471 υπέρ, ε, ψηφίζεται μάλλον. Δεκτή. 472 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 473 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 473. Τέλος. Παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια σας. 474 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 474. Τέλος. Δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική τι ταφ Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε στην ΤΕΒΕ 37. 479. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχω ηλεκτρονικά. Δεν είναι σαφές. «31 υπέρ 25 κατά εγκρίνεται». «84 υπέρ». «Κατά». «Αποχές». Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Το καταλαβαίνω γιατί είναι μακρά η ψηφοφορία, αλλά πρέπει να σηκώνετε τα χέρια. Λοιπόν, 84 ηλεκτρονικά. Πέρας. ...37 υπέρ, 20 κατά. Με μεγάλη διαφορά. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο όταν δεν τα χέρια σας. 85 η επόμενη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ντεβε 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύε 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 480 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 481 υπέρ. Κατά. Αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Την 481. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ 29 κατά απορρίπτεται συμβιβαστική U, λατινικό ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τι γίνεται. Δεν σας άκουσα. «493 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». Να σας υπενθυμίσω ότι για 10 λεπτά ακόμη, 10-12 λεπτά ακόμη θα έχουμε διερμηνία και πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ολοκληρώσει, αλλιώς θα, θα συνεχίσουμε χωρίς διερμηνία. Ντέβε 40, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 494 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε, ναι, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Might be. 27 uh, υπέρ 29 κατά. Απορρίπτεται. 495 η επόμενη ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 496 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 497 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 498 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 499-88 από κοινού ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 500 ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 501 ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 502 ψηφιπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Εντάξει. Πέρασε. 23 ψήφοι υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται επομένως 503 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 504 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 505 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική β λατινικό ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται που πηγαίνουμε στην 515 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Πέρες. 24 υπέρ 29 κατά, επομένως απορρίπτεται. 516 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 516. Πέρας. 32 ψήφοι πέρα, εγκρίνεται. Μόνο 22, 21 ήταν οι ψήφοι οι αντίθετες. Ε, 447 υπέρ, κατά, μάλλον 517. Η 447 τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 520 υπέρ, Την 519 την ψηφίσαμε με τη 244. 520 τώρα ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 521. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 522. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στα παραρτήματα. 523 υπέρ. και 524. Έχετε, δίκιο. Υπέρ, σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Χέρια. 525 και 526 τώρα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 527, 530, ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 528 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 529 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 529. 30 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 531 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Προσπαθήστε να παρακολουθείτε την ψηφοφορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε τι γίνεται. Πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 532. Ναι, είναι σαφές, αλλά πολύ λιγότερα χέρια σηκώνονται. 532 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 533 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 και 42 Θέλετε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 533. Αλλά επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας. Πέρασε. «33 υπέρ 21 κατά» η ψήφη. 92 και ντεβε 42 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ντεβε 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 534 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Πώς ε, Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 32 υπέρ 20 κατά. 535. 535 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 536 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στις 539 και 540 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 542 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιούρι 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 544 είναι η επόμενη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται συμβιβαστική W. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις ετουλικές αναφορές, τα citations, 94 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, 95 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, 96 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται, 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική X στις ετολικές σκέψεις recitals υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 23 κατά. Άρα εγκρίνεται. 101 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κα, ε, συγγνώμη, 2. 2 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Η διερμηνία διακόπτεται. Against, abstention adopted. 103 in favor. Against, abstention adopted. Deve 2 in favor. Against, abstention adopted. Deve 3 in favor. Against,